Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας και καλωσορίζω και ευχαριστώ όλος ιδιαιτέρως ε, τους αντιπροέδρους Σασόλη και Βίλαντ που πάντα ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις μας ε, για να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας όταν συζητάμε τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ και χαιρετίζω τον κύριο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βέλεν. Ο συγκεκριτής μας είναι ο κύριος Ρίμπιχ. Όπως θα έχετε διαπιστώσει, είμαστε στη συνήθεια διαδικασία. Ε, υπήρξε ένα σχέδιο για την μεταρρύθμιση της ε, δημοσιονομικής διαδικασίας, αλλά η Σοφή είπαν ότι θα πρέπει να παγώσει και ενδεχομένω να βγει από το ψυγείο μετά τι επόμενε ευρωεκλογέ. Άρα δεν είναι η συνήθι κατάσταση, αλλά είναι ε, η επαναφορά στη συνήθι διαδικασία. Λοιπόν, πρώτα στον κύριο Ρούμπι θα δώσω το λόγο για μία σύντομη εισαγωγή. Και κατόπιν οι αντιπρόεδροι όλοι και Βίλαντ θα πάρουν το λόγο. Και ο Γενικός Γραμματέας επίσης θα πάρει το λόγο. Ο κύριος Ρούμπιχ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο κύριο Αρτουή. Είμαστε τώρα σε μια σημαντική φάση. Έχουμε τους αντιπροέδρους μας, τους γνωρίζουμε πολύ καλά. Δεν είναι η πρώτη συζήτηση μαζί τους. Έχει διαμορφωθεί μια παράδοση για τη συζήτηση και χαίρομαι ιδιαίτερα που και οι σκιώδεις ε, γνωρίζουν τη διαδικασία. Δεν θα πω ότι είναι η συνήθιση διαδικασία γιατί υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Ο προϋπολογισμός του 19 δεν είναι ο συνήθις. Έχουμε δύο σημαντικά θέματα. Το ένα είναι βεβαίως ε, έτος εκλογών. Άρα υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Θα υπάρξουν λοιπόν κάποιες ιδιαίτερες δαπάνες. Για μας είναι πολύ σημαντικό να αυξηθεί η συμμετοχή στις ευρωεκλογέ. Αυτή είναι η πραγματική μας νομιμοποίηση. Εάν επαναληφθεί η κατάσταση του 2014, όπου στη Σλοβακία για παράδειγμα ψήφισαν μόνο το 13%, αυτό θα ήταν ιδιαίτερα επιζήμιο. Θέλουμε να αυξηθεί η συμμετοχή στις εκλογές. Και αυτό χρειάζεται τις αναγκαίες πιστώσεις. Και ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα, κύριο Βέλε, που εδώ και πολλά χρόνια, όταν προκύπτει έτος εκλογών, μα στηρίζει πάντα. Και η υπηρεσία ερευνών μας θα πρέπει να κάνει περισσότερα. Να μας δώσει ειδική πληροφόρηση, να μας δώσει στοιχεία ελεγμένα, που να μπορέσουν να αξιοποιηθούν από, άλλες τις πολιτικές, από όλες τις πολιτικές ομάδες και για να αντιμετωπίσουμε και τις ψεύτικες ειδήσει, τα fake news, ούτω ώστε να ενημερωθούν ε, για τέτοια ενδεχόμενα οι βουλευτές και για να αποδείξουμε ότι το Κοινοβούλιο εργάζεται σοβαρά. Και γι' αυτό κάναμε και τις αντίστοιχες εκδηλώσεις στο Στρασβούργο. Γιατί διαπιστώσαμε ότι με μεγάλη καθυστέρηση και ανεπαρκώς επανειλημμένα έχουμε αντιδράσει σε κάποια τέτοια fake news γιατί δεν ενημερωθήκαμε έγκαιρα. Και μετά διαπιστώνουμε ας πούμε σε όλες τις εφημερίδες ε, της Ευρώπης και σε όλες τις τηλεοράσεις να λέγονται πράγματα τα οποία μετά πρέπει να διευκρινίσουμε μετά από δύο-τρεις μέρες ότι δεν ισχύουν. Πρέπει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρουσιάσει στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών πρέπει να έχουμε μια επικοινωνιακή στρατηγική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να κάνουμε μια συζήτηση και να κερδίσουμε τη συζήτηση για το μέλλον της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Να μην ξεχνάμε ότι στην ε, Μεγάλη Βρετανία το 1 τρίτο των ψηφοφόρων αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, να μην συμμετέχουν πλέον στο ίδιο τραπέζι με εμά στη λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι λυπηρό. Επανερχόμεθα σε διακρατικές σχέσεις που στο παρελθόν ε, έχουν δημιουργήσει τεράστιες ζημιές. Πρέπει λοιπόν να προβάλλουμε τη δημοκρατική φύση των, ευρωπαϊκών θεσμών και να αντιμετωπίσουμε τους στρατούς από τρόλ που περιμένουν εκτός Ευρώπης για να συμμετάσχουν στις, ε, στην προεκλογική εκστρατεία. Άρα βεβαίως χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό, προσωπικό που να έχει τις ανάλογες γλωσσικές γνώσεις. Το δεύτερο, πέρα από την επίσημη επικοινωνιακή στρατηγική του Κοινοβουλίου, είναι σημαντικό και τα πολιτικά κόμματα να μπορέσουν να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους. και να δώσουν στους ε, ψηφοφόρους τη δυνατότητα να επιλέξουν με βάση τις απόψεις για διαφορετικά θέματα των διαφόρων πολιτικών ε, κομμάτων. Βεβαίως ε, έχουμε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών δυνάμεων που συμμετέχουν. Κανένα κοινοβούλιο στον κόσμο δεν έχει τόσο ευρεία πολιτική εκπροσώπηση. Και όποιος παρακολουθεί την καθημερινή μας εργασία θα διαπιστώσει ότι είμαστε επίσης ένα κοινοβούλιο το οποίο συζητάει για τόσο πολλά θέματα σε τόσο μεγάλο βάθος. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό και τα πολιτικά κόμματα που έχουν ε, διαφορετικές απόψεις να έχουν δυνατότητα να τις παρουσιάσουν, ούτως ώστε κάθε ψηφοφόρος να αποφασίσει ε, πώς θα ψηφίσει, ποιος εκπροσωπεί καλύτερα τα συμφέροντά του. Και η πολιτική δουλειά των κομμάτων είναι σημαντική. Ξέρουμε όλοι ότι τα κόμματά μας στα κράτη μας δεν είναι πραγματικά διατεθειμένα να κάνουν μια προληπτική εκστρατεία που να αναφέρεται κυρίως στην Ευρώπη. Θυμάμαι, όταν πέρασα από την τομική οργάνωση στην ε, περιφερειακή οργάνωση, στην εθνική οργάνωση, ο καθένας έλεγε σε κάθε επίπεδο, ο καθένας ασχολείται περισσότερο με τα δικά του. Πρέπει λοιπόν να προβάλλουμε τα ευρωπαϊκά κόμματα και να μπορέσουμε να τους δώσουμε και τα αναγκαία μέσα, τους αναγκαίους πόρους. Επίσης, έχουμε το γεγονός ότι γύρω στο 50% θα αποχωρήσουν, των συναδέλφων θα αποχωρήσουν από το Κοινοβούλιο. Άρα χρειάζονται κάποιες μεταβατικές ε, πληρωμές, όχι μόνο για τους αποχωρούντες συναδέλφους, αλλά και για τους βοηθούς τους. Και επίσης και για τους ε, μαθητευόμενους. Ελπίζουμε να εφαρμοστεί τώρα το τελευταίο τμήμα της χρηματοδότησης για αυτούς τους αποχωρούντες. Αυτές είναι οι σημαντικές μας προτεραιότητες. Για μένα και τους κοσμήτορες το σημαντικό είναι το ερχόμενο κοινοβούλιο να είναι σε θέση να ε, κάνει τη δουλειά του με αξιοπρεπείς συνθήκες, με ε, επαρκή γραφεία, επαρκή και σύγχρονο εξοπλισμό. Και βεβαίως να μην ξεχάσουμε ότι θα έρθουν πολλοί νεότεροι συνάδελφοι που θα έχουν πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις από την πληροφορική και τις υπόλοιπες δυνατότητες εξοπλισμού που θα πρέπει να τους προσφέρει το σώμα και για την επικοινωνιακή τους πολιτική Πρέπει λοιπόν να έχουμε το 1 συν 2 γραφεία στις Βρυξέλλες και το 1 συν 1 γραφεία στο Στρασβούργο. Και θα πρέπει να υπάρξουν και μέτρα επιμόρφωσης, όχι μόνο για τους νέους συναδέλφους, αλλά και για τους βοηθούς τους, που θα είναι και αυτοί νέοι. Και θα πρέπει να δούμε <clears throat> εάν κάποιοι υπάλληλοι των πολιτικών ομάδων να ε, περάσουν σε καθήκοντα βοήθειας προς τους βουλευτές. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν και εκεί οι αναγκαίες προσαρμογές της ε, γιατί ένας συνεργάτης της ομάδας ε, γίνεται συνεργάτης βουλευτή, αναμένει να έχει τα κατάλληλα κίνητρα για να επιχειρήσει αυτή την αλλαγή. Έχει έννοια λοιπόν να το κάνουμε και αυτό. Τελευταίο. Συνεχίζεται η εργασία για την ασφάλεια κυρίως για το κτίριο ΚΑΝΤ και τις μεταφορές από και πρών. Το Κοινοβούλιο μπορεί να αυξήσει την ε, αποτελεσματικότητά του στον τομέα αυτό και ελπίζω να γίνουν τα απαραίτητα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εισαγωγή. Τώρα θα δώσουμε το λόγο ε, στους αντιπροέδρους. Ποιος θέλει πρώτος να πάρει το λόγο. Ο κύριος Ασολή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Ρούμπιχ. Μαζί συνεργαστήκαμε και με εσά βεβαίω. Ε, συνεργαστήκαμε στους προηγούμενους ε, προϋπολογισμούς. είμαστε πολύ εξασκημένοι, πολύ προπονημένοι σε αυτή την διαλεκτική άσκηση, διανοητική άσκηση. Ο προϋπολογισμός του 2019, όπως είπε και ο κύριος Ρούμπιχ, είναι μια διαφορετική άσκηση από τις προηγούμενες. Γιατί είναι χρονιά εκλογική και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μια σειρά από ερωτήσεις και προβλήματα που δεν είχαμε στους προηγούμενους ε, προϋπολογισμούς. Αυτό δεν θα πρέπει να μας ε, προκαλέσει κανένα πρόβλημα, γιατί αυτό που πρέπει να κάνουμε πάνω απ' όλα είναι να λειτουργεί σωστά και χρηστά ο οίκος μας. Το 2019 βεβαίως θα έχουμε κάποια έκτακτα έξοδα που είναι ίδια μιας εκλογικής χρονιάς γιατί έχουμε τα, τις δαπάνες ε, του τέλους της εντολής, ε, έχουμε τις αποζημιώσεις των ε, βουλευτών που θα φύγουν από το Κοινοβούλιο, επίσης αποζημιώσεις για βοηθούς οι οποίοι θα λήξουν η σύμβασή τους και δεν θα συνεχίσουν να δουλεύουν για το Κοινοβούλιο. Έχουμε επίσης τα έξοδα για την προεκλογική εκστρατεία, που όπως είπε ο κύριος Ρούμπιχ είναι πολύ σημαντικά. Αυτές οι γραμμές του προϋπολογισμού είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, είναι η μερίδα του, λέ, του λέοντος των εκτάκτων εξόδων. Συνολικά η κατάσταση μας οδηγεί σε αύξηση του προϋπολογισμού για το 2019 κατά 3,9% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2018. Παρ' όλα αυτά, θα πάρουμε το 18,8% του 20% που θα έπρεπε να πάρει το Κοινοβούλιο από την πέμπτη γραμμή, διοικητικά έξοδα δηλαδή, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Παίρνουμε λοιπόν το 18,8% από το 20% και ποσοστιαία αυτό είναι το χαμηλότερο ποσοστό τα τελευταία 15 χρόνια η διαπραγμάτευση μεταξύ της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου για την έξοδο του δεύτερου από το Ηνωμένο Βασιλείο μας οδήγησε σε μια συμφωνία ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετάσχει στους προϋπολογισμούς 2019 και 2020. Το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2019 λαμβάνει υπόψη ότι θα έχει το Κοινοβούλιο 700 51 ευρωβουλευτές και 28 χώρες, χωρίς να εξετάζουμε αυτή τη στιγμή την έκθεση πρωτοβουλίας στην Επιτροπή ΑΦΚΟ για τη σύνθεση του Κοινοβουλίου που τη στιγμή που η Μεγάλη Βρετανία θα φύγει από την Ευρώπη θα σημάνει και μείωση των ευρωβουλευτών στους 705. Λοιπόν, αποζημίωση θα πρέπει να, να, ε, να δώσουμε αυτή την αποζημίωση στους ε, ευρωβουλευτές που δεν θα ξανά είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς και στους βοηθούς τους για την ε, καταγγελία της σύμβασής τους ή την απόλυσή τους. Επίσης, διάφορες δαπάνες λόγω του τέλους της θητείας μας που αναφέρονται λεπτομερώς στο σχέδιο προϋπολογισμού που θα λάβετε, θα λάβετε προεκλογική εκστρατεία. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για το Κοινοβούλιο και θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε, αντιμετωπίσουμε μια τάση αντιευρωπαϊκή πολύ έντονη. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε προσπάθεια σε πολλά επίπεδα για να ενημερώσουμε τον κόσμο και να δράσουμε ε, απέναντι σε εκείνες τις κατηγορίες ε, των Ευρωπαίων πολιτών που μπορεί να τους ενδιαφέρει το ευρωπαϊκό project αλλά που θα πρέπει όμως να πάνε να ψηφίσουν, γιατί μπορεί να μην θέλουν να πάνε να ψηφίσουν ή να βαριούνται για οποιονδήποτε λόγο. Ε, και αυτοί θα, είναι, θα αντιπαρατεθούν στους ε, εχθρικούς προς, το, προς την Ευρώπη ψηφοφόρους. Επίσης, μην ξεχνάτε τις συζητήσει που, γίνεται, που γίνονται στο, για το Brexit αυτέ αυτές τις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη, άρα θα πρέπει η εκστρατεία μα να είναι σε πολλά επίπεδα, θα πρέπει να γίνει ε, σε πολλού τομεί σε, με τα πολιτικά κόμματα και με το Κοινοβούλιο. Το 2019 έχουμε προβλέψει 8,3 εκατομμύρια ευρώ που θα προσθεθούν στα 25 εκατομμύρια του 2018. Γιατί ήδη από πέρυσι Είχαμε προβλέψει ένα ποσό για την προεκλογική εκστρατεία. Έτσι. Έχουμε λοιπόν 8,3 εκατομμύρια επιπροσθέτω στον 25 που είχαμε, το, που είχαμε προβλέψει το 18. Επειδή ακριβώς ε, θα κάνουμε αυτή την ε, πολυμέτωπη προσπάθεια, τον πολυμέτωπο αγώνα, αγώνα θα έχουμε τον Spitzenkandidaten για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι νομίζω σημαντικό να δώσουμε την δυνατότητα στα ευρωπαϊκά ε, πολιτικά κόμματα να έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν την προεκλογική εκστρατεία εξοπλισμένη. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Παράλληλα, είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την προσπάθεια επικοινωνίας προς τα γραφ... δηλαδή να έχουμε μια επαφή με τα γραφεία του Κοινοβουλίου στις χώρες μας, για να έχουμε μια πιο άμεση επαφή με τις χώρες. Προβλήματα ασφάλειας. Όπως ξέρετε, εδώ και χρόνια ο... οι προπολογισμοί μας προβλέπουν παρεμβάσεις για λεπτά ευαίσθητα θέματα που ανακάλυψε το Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή στέθηκε ψηλά στην ατζέντα μας με δραματικό τρόπο το θέμα της ασφάλειας. Που από τότε που η τρομοκρατία χτύπησε την πόλη των Βρυξελών. Έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις συγκεκριμένες. Η πρώτη είναι να ολοκληρώσουμε την, τα έργα στην είσοδο Vice για να είναι ασφαλής αυτή η είσοδος, να ολοκληρώσουμε και τα έργα στα άλλα κτίρια Μιλάμε για έργα που έχουν ξεκινήσει το 2016, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Για το 2019 προβλέπονται σημαντικές επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση, κυρίως για την είσοδο του κτηρίου ΒΑΙΣ και προβλέπεται να φτιάξουμε μια δομή για να έχουμε και μια υποδοχή για τους επισκέπτες και ένα παβίλιο, ας πούμε, ένα χώρο για το, τους ελέγχους ασφάλειας. Αυτό μου φαίνεται πολύ ωραίο. Σχέδιο ε, έργο IPAX. Το εγκρίναμε στο Προεδρείο του 2015 με τις πρώτες επιθέσεις στο Παρίσι. Το... Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να έχει μια τεχνολογία για την ασφάλεια εντελώς ε, μοντέρνα. Φυσικά είναι ένα σύστημα το οποίο θα βελτιώσει την ασφάλεια της ε, πρόσβασης στο Κοινοβούλιο. Θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε το προσωπικό ασφαλείας και να μας κάνει και θα μας εξασφαλίσει και η οικονομία για να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε απαρχαιωμένη τεχνολογία. Πάντα για το θέμα της ασφάλειας, ένα βασικότατο θέμα είναι η ασφάλεια στην πληροφορική. Υπάρχει ένας υπεύθυνος εδώ και ένα χρόνο για την ασφάλεια. Είναι υπεύθυνο για όλα αυτά τα θέματα, για τις απειλές στην πληροφορική κτλ. και αυτή η θέση θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, γιατί ξέρετε ότι η ασφάλεια στην πληροφορική θα εξακολουθεί να είναι ψηλά στην ατζέντα, γιατί θα υπάρχουν συνεχώς επιθέσεις στην πληροφορική. Λοιπόν, για τα κτίρια, να βελτιώσουμε το χώρο εργασίας των βουλευτών και βοηθών. Αυτό δεν είναι προαιρετικό, είναι ανάγκη. Μια και είναι όπως είναι τα γραφεία μας, είναι αυτό που θα κληροδοτήσουμε στους επόμενους βουλευτές. Ε, θα πρέπει να το κληροδοτήσουμε σε καλή κατάσταση και σε, να το βελτιώσουμε. Για το 2019 επίσης θα έχουμε project μονο, μονοετή και πολυετή. Το 2019 θα πρέπει το κτίριο ΚΑΝΤ στο Λουξεμβούργο, στην, η ανατολική του πτέρυγα να ολοκληρωθεί. Θα συνεχιστεί το e-Parliament, αυτό το project που είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό, ούτως ώστε και οι συνεργάτες μας και εμείς και οι διοικητικοί πάλι να έχουμε τη δυνατότητα κάποιων μοντέρνων εργαλείων για τις εργασίες μας και να προσφέρουμε νομοθετικές υπηρεσίες και ε, κοινοβουλευτικές ε, υπηρεσίες ακόμα καλύτερες. Τελευταίας τεχνολογίας. Είναι χρήσιμο το project ERMS για τη διαχείριση των εγγράφων ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλος, τελευταία παρατήρηση για τον προϋπολογισμό τελευταία ενημέρωση καλύτερα, όχι παρατήρηση, η μείωση του προσωπικού. Για να φτάσουμε στο 5% της μείωσης του προσωπικού, όπως είχαμε συμφωνήσει με βάση την διαθεσμική συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα χάσει 59 θέσεις. Παρατείναμε κατά ένα χρόνο αυτή την απόφαση για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο του 5% και ελπίζω πραγματικά να μην μας ζητήσει, να μην μας ζητήσει κανένας να κάνουμε επιπλέον προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί έχουμε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει στα πλαίσια της Διαθεσμικής Συμφωνίας. Το Κοινοβούλιο έκανε σημαντικότατες προσπάθειες, ήταν το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο, το οποίο τιμωρήθηκε πιο πολύ από, από οποιοδήποτε άλλο, από τη μείωση του προσωπικού. Εμείς σεβαστήκαμε τις δεσμεύσεις μας και θα πρέπει να μας αναγνωριστεί αυτό. Ευχαριστώ. Merci, merci, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Ο Αντιπρόεδρος Βίλαντ έχει το λόγο τώρα. Ja, vielen Dank, Herr äh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ορισμένα υπόθηκαν. Εγώ θέλω να τονίσω και επισήμως ότι για τα θέματα και της ε, απτής ασφάλειας αλλά και της κύβερνο ασφάλειας ορισμένα είναι ακόμη στην αρχή. Οπότε θα χρειαστεί να κάνουμε πολύ περισσότερα στο μέλλον. Στην πληροφορική γενικώ πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της διασυνδεσιμότητας ε, σε ένα σύγχρονο κόσμο. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα ακόμη γι' αυτό. Ο προπολογισμό μας βεβαίως προβλέπει, αν το δει κανείς σε πρώτη ανάγνωση, 3,9% αύξηση που φαίνεται μεγάλη βέβαια. Αλλά αν δούμε τις δαπάνες λόγω των εκλογών που είναι 1,2% της αύξησης, το 1,2 από το 3,9 αυτό, αλλά θέλω να διευκρινίσω ακόμη περισσότερο. ότι θα πάρουμε το 18,79% των δαπανών της κατηγορίας 5. Είναι το χαμηλότερο ποσοστό της τελευταίας πενταετίας. Και δεν εξαντλεί το 20%. Μας δίνει λοιπόν ένα περιθώριο 130 εκατομμυρίων. 1,2% δηλαδή των δαπανών της ε, κατηγορίας 5 είναι 130 εκατομμύρια, τα οποία δεν θα ζητήσει το Κοινοβούλιο. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε και στο μέλλον περισσότερο. Το 49 ε, σημείο των ε, κειμένων που έχετε μπροστά σας ε, αναφέρονται στα θέματα των γραφείων του βουλευτέ, ένα συν δύο Βρυξέλλε, ένα και ένα στι Βρυξέλλε, στο σημείο 55, βλέπετε, κάτι που θεωρώ ως το μεγαλύτερο ε, σημερινό έλλειμμα και που εγώ ε, θεωρώ προσωπικά ως την ε, μεγαλύτερη ήττα μου στη σημερινή μου δραστηριότητα αφορά την ανακαίνιση του κτηρίου Πολαρή Σπακ που δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν και όλοι ξέρουν ότι είμαστε σε μια ιδιαίτερα επισφαλή κατάσταση. Δεν είναι μόνο προσωπική τα για μένα. Αυτό είναι ανεπάρκεια και της εργασίας του Προεδρείου και όλων όσων ασχολούνται με αυτά τα θέματα στο σώμα. Θα οδηγηθούμε αντικειμενικά σε μια κατάσταση που ε, θα είναι πολύ δύσκολο κατόπιν να ανατραπεί. Στα σημεία 49 και 57 θα δείτε ε, αυτά που προτείνουμε για το θέμα η ευρωπαϊκή εμπειρία. Και εδώ η κατάσταση είναι ευάλωτη του προπολογισμού. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα. Ο πρώην πρόεδρος Σούλτς στο Βερολίνο είχε εκφραστεί ενθουσιοδός ε, ε, υπέρ του προγράμματος αυτού. Στο Στρασβούργο υπήρξαν μια σειρά από τέτοιε δραστηριότητε και για το κινηματογράφο 360 μοιρών και για τα παιχνίδια ρόλων. Ήταν ε, ενθουσιώδης η αντίδραση των συμμετεχόντων. Συζήτησα με το Βαβαρικό Υπουργείο Πολιτισμού και μου είπαν ότι αυτό το παιχνίδι ρόλων που μου είπε κύριε Βίλαν μόνο στο Ισραήλ υπάρχει κάτι το ανάλογο. Και στην πρώτη ομάδα, γιατί συμμετείχα και εγώ, σε αυτό το παιχνίδι ρόλων ως Πολωνός σοσιαλιστής ε, πήρα το λόγο, ναι βεβαίως πήρα το λόγο και καθόμουν μεταξύ των ε, συναδέλφων της πολιτικής ομάδας αυτής ο πρώτος νέος που μου μίλησε μου είπε κύριε Βίλαντ καταπληκτική δουλειά επιτέλους κάτι το οποίο μπορεί να καταλάβει η νεολαία μιλάτε στη γλώσσα της νεολαίας παίρνουν ένα smartphone οι νέοι λαμβάνουν ε, εντολές και η εργασία τους είναι ε, πολύ καλά πλαισιωμένη. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να δείτε πώς ε, λειτουργούν αυτά στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και σε διάφορες πρωτεύουσες. Και ευχαριστώ πολύ τον Γενικό Γραμματέα και τη Γενική Διεύθυνση που το οργάνωσε. Τώρα για το οργανόγραμμα. 79 και επόμενα σημεία. Νομίζω ότι ήδη φτάσαμε στο όριο και δεν πρέπει να το υπερβούμε της μείωσης θέσεων. Δεν θα σήμαινε βελτίωση. Εντάξει, μπορεί να μειώναμε περισσότερο τις δαπάνες προσωπικού, αλλά θα είχαμε πλέον αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του σώματος. Και δεν θα θεωρούσα μελλοντικές συμφωνίες επί ποσοστών μειώσεως ως θετικές, γιατί ξέρω ότι η Κομισιόν μπορεί να κάνει διάφορα κόλπα, να στείλει προσωπικό στους αποκεντρωμένους οργανισμούς και το Συμβούλιο έχει απεριόριστους πόρους στην ουσία στη διάθεσή του από τα κράτη-μέλη. Ξέρω ότι πολλοί λένε διάφορα Υπάρχουν ομάδε επισκεπτών και πολλοί μου λένε Μα πώ εργάζονται εδώ μέσα. Και εγώ του λέω. Δεν ξέρω, εγώ τους απαντάω, δεν ξέρω πώς καταλαβαίνουν αυτή την ε, απάντηση. του λέω 50%. Αλλά τονίζω ότι οι εργαζόμενοι μας δουλεύουν πολύ σωστά. Τώρα για το θέμα των γλωσσών. Θέλω να είμαι ιδιαίτερα κατηγορηματικός γι' αυτό. Όταν θα φύγει η Βρετανία, φυσικά τα αγγλικά μέχρι στιγμής εκπροσωπούνται στο σώμα και υπήρχαν ως γλώσσα εργασία και πριν την είσοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε όλοι. Αν δείτε εδώ πώς είναι η σειρά των γλωσσών, εδώ πώς είναι οι καμπίνες. εκπροσωπούν τις ομάδες χωρών όπως εντάχθηκαν στην Ένωση. Οι πρώτες πέντε γλώσσες είναι γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά. Μετά έχουμε τις πρώτες χώρες διεύρυνσης και στο τέλος έχουμε τις ε, νέες ε, γλώσσες των χωρών που μπήκαν το 2004 και το 2007. Τα αγγλικά ήταν από την αρχή γλώσσα εργασίας εδώ. Και είναι γλώσσα που εφαρμόζεται, που ε, είναι χρήσιμη σε όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε, στους 200, για τα 200 εκατομμύρια Νιγηριανών δεν τα εξυπηρετεί πάρα πολύ που η γλώσσα τους είναι η μεγαλύτερη μετρική γλώσσα στον κόσμο, εάν δεν τη μιλάει κανένας άλλος. Άρα, με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, κανείς, εάν αυτό θα σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να μιλάει πια τη γλώσσα του, γι' αυτό θα πρέπει να το θεωρήσουμε πλεονέκτημα το ότι θα διατηρηθούν τα αγγλικά. Λοιπόν, 3,9% αύξηση. Το κοινοβούλιο μας ε, δαπανά 4 ευρώ ανά πολίτη. Το αμερικανικό σύστημα κοστίζει 5 εκατομμύρια στον κάθε πολίτη. Παρά το ότι το αμερικανικό σύστημα έχει δεν έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των δύο διαφορετικών εδρών, 150 εκατομμύρια, ούτε την πολυγλωσία, που μα κοστίζει περίπου 450 εκατομμύρια. Δηλαδή ένα τρίτο περίπου του προπολογισμού μα, προλογισμού μας αφορά κόστος για το οποίο δεν φέρουμε καμία ευθύνη εμείς. Και για ένα κόστος το οποίο δεν αφορά τους Αμερικανούς. Δηλαδή, στην ουσία, αναπολίτη κοστίζουμε περίπου τα μισά από ό,τι τους Αμερικανούς. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να αυτομαστιγωνόμαστε. Θα πρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί και επιθετικοί. Λοιπόν, τα προβλήματα λοιπόν αφορούν κυρίως ε, τα κτίρια. Θα πρέπει για την κτηριακή πολιτική να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί, να έχουμε ένα μητρό χώρων. Όταν ο συνάδελφος ε, Ντεπρέν στο Στρασβούργο θα πρέπει να υπάρχουν ευφύης εφαρμογές που να ξέρουν ότι είναι στο Στρασβούργο. Και αυτές τις μέρες να μην πηγαίνει καθαρίστρια στο γραφείο του. Υπάρχουν σύγχρονες δυνατότητες που μπορούν να διευκολύνουν την κατάσταση, δηλαδή ε, να ε, μην παρέχονται ορισμένες υπηρεσίες όταν δεν χρειάζονται. Έχουμε λοιπόν ακόμη περιθώριο για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας. Θα πρέπει και οι επιτροπές να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους, γιατί οι επιτροπές από μόνες τους αποφασίζουν αν θα κάνουν άλλη μία αποστολή fact-finding ή αν θα ακούσουν άλλον έναν εμπειρογνώμονα ή ε, αν εδώ θα υπάρχουν δύο μπουκάλια νερό για τον πρόεδρο θα πρέπει να αναλάβουν περισσότερη ευθύνη. Για να υπάρχει πιο υπεύθυνη ε, χρήση των πιστώσεων. Αυτό αφορά και τις συνεδριάσεις ε, των επιτροπών στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, συγγνώμη και αφορά και τι Ολομέλειε εδώ στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες έχουμε πολλές συνεδριάσεις που δεν είναι απαραίτητες και αν θέλουμε να κάνουμε εξοικονομήσεις τότε μπορούμε πραγματικά να μειώσουμε τις πατάλες. Και αν κάποιο δεν είναι τακτικό μέλο μια επιτροπή, δεν είμαι σίγουρο ότι χρειάζεται να κάνει τροπολογίε. Για κάτι ακόμη, αυτή τη βδομάδα και σα καλώ ευχαρίστω όλου, ε, κάνουμε νέα πράγματα σε πέντε τομείς δραστηριότητας. Πρώτα απ' όλα είπαμε ότι δεν χρειαζόμαστε νέα έπιπλα. Επίσης, η επιδιόρθωση μέσω υπεργολαβίας μας κοστίζει όλο και περισσότερο. Οι επιστήμονες ασχολούνται με το θέμα του σύγχρονου εξοπλισμού. Κάθε 20 χρόνια πρέπει να ανακαινίζεται πλήρως εξοπλισμός ή θα πρέπει να γίνονται κάποιες ε, εναλλακτικές χρήσεις. Και επίσης έγινε μία προκήρυξη και έχουμε πέντε που συμμετέχουν σε αυτή την προκήρυξη με τους οποίους συζητάμε. Τους προτείναμε να μας πούν, να μας κάνουν μια πρόταση για το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί το γραφείο του βουλευτού, του κάθε βουλευτή, η χώρη αναμονή. η Σασόλη, Μωαγάν Σαρτιέ, Λιμπεράσκη, Κάρσκη και εγώ, υποφαινόμενος, θα λάβουμε τέτοια πρότυπα γραφεία και θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν και καλό και τους συναδέλφους θα θέλουν να δουν πώς θα είναι αυτό το ε, πρότυπο γραφείο μου και του κυρίου Σασόλη, πώς θα είναι ο χώρος αναμονής για να ε, προσαρμόσουμε περισσότερο τα γραφεία μας στις ανάγκες των βουλευτών χωρίς όμως να ε, εγκαταλείψουμε και τις προσπάθειες περαιτέρω εξοικονομήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Βίλαντ. Να επισημάνω ότι η διερμηνία θα έχουμε μέχρι τις 6.30. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος να συνεχίσουμε στα αγγλικά. Κύριε Γενική Γραμματέα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι αντιπρόεδροι ήδη ε, αναφέρθηκαν σε πολλά θέματα. Θα αναφερθώ μόνο σε θέματα τα οποία δεν έχουν εξηγηθεί ε, αναλυτικά και λόγω της, ε, του περιορισμένου χρόνου. Βεβαίως υπάρχουν κάποια κάποιες αβεβαιότητες για τον προπολογισμό. Η πρώτη είναι το Brexit. Από το Δεκέμβρη ε, βεβαίως έχουμε την ε, ελπίδα ότι μέχρι τέλος του 20 θα είναι εγγυημένη η χρηματοδότηση, αλλά όλα σχετίζονται με όλα όπως πάντα λέγεται. Με την συμφωνία αποχώρησης, με τη μεταβατική περίοδο, με την μελλοντική σχέση. Αυτή τη στιγμή υποθέτουμε σε αυτή την πρόταση για τον προπολογισμό ότι για το πλαίσιο του, υπάρχον, του υπάρχοντος ΠΔΠ θα συνεχίσει να υπάρχει χρηματοδότηση. Αλλά δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε να υπάρξει κρίση διαπραγματεύσει. Οπότε θα πρέπει να γίνουν προσαρμογέ. Αλλά αυτό θα αφορά όλα τα θεσμικά όργανα. Και από ό,τι φαίνεται θα διορθωθεί με μια διορθωτική επιστολή, με μια τροποποιητική επιστολή. Αλλά υπάρχει αυτή η βεβαιότητα για τον προπολογισμό θα έχει βεβαίως τον Brexit και διοικητικέ επιπτώσεις. Ο Πρόεδρος παρακάλεσε σε μία από τις ε, ερχόμενες συνεδριάσεις του Προεδρείου το Φεβρουάριο από ό,τι φαίνεται λέει ο κύριος Γενικός Αματέας θα μιλήσουμε με τον Μισελ Μπαρνιέ και τον κύριο Φερχόφστατ παρακάλεσα τις γενικές διευθύνσεις να μου πούν πού θα τεθούν τα κυριότερα θέματα σε σχέση με τον Brexit και νομίζω ότι θα είναι κυρίως σε τέσσερις τομείς. Πρώτον, τι θα γίνει με τους Βρετανούς συνεργάτες μας. Δεύτερον, τι θα γίνει με τα αγγλικά αν θα εξακολουθήσουν να είναι γλώσσα εργασίας. Τρίτον, τι θα γίνει με τις προκηρύξεις. Θα δώσουμε μεγάλης διάστασης ε, και ευαίσθητα συμβόλαια στο μέλλον και εκτός της Ένωσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Ή όχι και τι θα γίνει με το γραφείο του Κοινοβουλίου. Το Προεδρείο έκανε μια πρώτη προκαταρκτική συζήτηση για τα θέματα αυτά, συζητώντας τον προπολογισμό για τους Βρετανούς υπαλλήλους μας. Ε, έχουμε 125 υπαλλήλους που έχουν μόνο βρετανική υπηκότητα. Τα δύο τρίτα είναι γλωσσικοί υπάλληλοι. Ξέρουμε ότι και στο μέλλον θα χρειαστούμε ε, αγγλόφωνους μεταφραστές και διερμηνείς και ε, ε, γλωσσομαθείς νομικούς και στον τομέα της επικοινωνίας. Αυτούς λοιπόν τους συνεργάτες θα συνεχίσουμε να τους χρειαζόμαστε βράχη και μέσο πρόθεσμα. Και για όλους τους υπαλλήλους ισχύει ότι δεν είναι απεσταλμένοι από τα κράτη-μέλη, είναι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή περισσότεροι σε σχέση με το μέσο όρο Βρετανοί είναι προχωρημένης ηλικία, πολλοί θα αποχωρήσουν ε, στο εγγύς Οπότε θα πρότεινα οι πάλι αυτοί, όχι μόνο οι γλωσσικοί αλλά και οι υπόλοιποι, να συνεχίσουν να εργάζονται για μας. Για τις γλώσσες μόνο ένα στοιχείο. 70% των τροπολογιών που υποβάλλονται στις επιτροπές υποβάλλονται στα αγγλικά. Βέβαια δεν τις ε, διατυπώνουν μόνο Βρετανοί, πάρα πολλοί βουλευτές που μπορούν να συντάσσουν στα αγγλικά. Άρα είναι σαφές ότι βράχει και μέσο πρόθεσμα δεν μπορούμε να καταλήψουμε τα αγγλικά. Για τα εξωτερικά γραφεία, τα γραφεία συνδέσμου όπως λέγονται, το Προεδρείο είπε μα έχουμε γραφείο στη Washington η μελλοντική μας σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο όταν θα αποχωρήσει σίγουρα θα είναι τουλάχιστον εξίσου στενή όσο η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχει ληφθεί απόφαση, αλλά η πρώτη τάση θα ήταν να πούμε ότι αυτό το γραφείο του Κοινοβουλίου στο Λονδίνο και στο Εδιμβούργο θα πρέπει να διατηρηθούν. Υποθέτω ότι το Προεδρείο θα αποφασίσει ενδεχομένως τη συνεδρίαση ήδη τον Απρίλιο που θα έχει και δημοσιονομικές επιπτώσεις λοιπόν και για τον προπολογισμό του 19. Ο κύριος Βίλαντ αναφέρθηκε ήδη στην κτηριακή πολιτική. Είναι σαφές ότι ε, έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την ε, κτηριακή πολιτική. Έχουμε επαρκές ε, επαρκή αριθμό γραφείων στο Στρασβούργο με το κτίριο Χάβελ. Τώρα εν ώψη των ευρωεκλογών ε, του 19 υπάρχουν διαφορετικές προτεραιότητες και στο Λουξεμβούργο. Είμαστε ε, μετά από πολύ χρόνο σε φάση επίλυσης των προβλημάτων με το κτίριο και στις Βρυξέλλες με τα εγκαίνια του κτίριου Μάρτεν στην 1η Απριλίου και με το κτίριο στην πλατεία Ντεμέους θεωρώ ότι οι ανάγκες μας έχουν καλυφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή πρέπει τώρα να διατυπώσουμε νέες προτεραιότητες. Και η ομάδα εργασίας ε, κτηριακή πολιτική στην επόμενη συνεδρίασή της, την επόμενη εβδομάδα, θα ασχοληθεί σε βάθος με τα θέματα αυτά, κατά τη γνώμη μου. Χρειαζόμαστε περισσότερους χώρους για τριμερείς διαλόγους. Όταν χτίστηκαν τα κτίρια αυτά, πριν περίπου 20 χρόνια δεν ε, υπήρχαν ε, τριμερείς διάλογοι. Σήμερα ένα τμήμα πολύ ουσιώδες της δουλειάς μας γίνεται μέσω των τριμερών διαλόγων. Για φέτος θεωρούμε ότι και προβλέπουμε 800 τριμερείς διαλόγους. Αλλά έχουμε μόνο τέσσερις αίθουσες ε, κατάλληλες. Και ορισμένες είναι μάλιστα και εν μέρη κατάλληλες. Άρα Πρώτο θέμα της μελλοντικής ε, κτηριακής πολιτικής θα είναι περισσότεροι χώροι για τους τριμερείς διαλόγου, διαλόγους. Δεύτερον, ε, θα θέλουμε να κάνουμε περισσότερα για το εμπειρία Ευρώπη. Οι πρώτες εμπειρίες που κάναμε ιδιαίτερα στο Βερολίνο, στο Στρασβούργο, αλλά και στη Λιουμπλιάνα ήταν πολύ θετικές. Από τότε που άνοιξε αυτή η δυνατότητα στο Βερολίνο την έχουν επισκεφθεί 250.000. Νομίζω ότι ε, μπορούμε να ε, ε, επικοινωνήσουμε με πολλούς πολίτες με λίγες δαπάνες και τη συμμετοχή λίγου προσωπικού και γι' αυτό αποφασίστηκε από την Επιτροπή Προϋπολογισμών να χρηματοδοτηθεί αυτό και από το Προεδρείο αποφασίστηκε να γίνουν περιορισμένα στο Ελσίνκι και στο Τάλιν. Εάν υπάρξει θέληση, τότε θα πρέπει να ε, γίνουν περισσότερα γι' αυτό. Επίσης, έχουμε το κτίριο ΤΡΕΒ 2. Γιατί ξέρετε ότι συνδέονται όλα μας τα κτίρια στις Βρυξέλλες. Θα μπορούσαμε, όπως λέει και η, ε, η Αστερίξ και ο Βελίξ, να πούμε ότι όλα μας ανήκουν εκτός από κάτι λίγο. Το κτίριο αυτό ανήκει στο Βελγικό Γραφείο Οικογενειακών Ασφαλίσεων. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει. Γιατί αυτή η υπηρεσία θα μετατραπεί σε περιφερειακή υπηρεσία. Επίσης πρέπει να γίνουν ανακαινήσεις κτίριων. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι και για περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς ε, λόγους κάθε χρόνο ένα 3% των κτηρίων μας που είναι σε κατάσταση που δεν είναι επαρκής από αυτή την άποψη θα πρέπει να ανακαινίζονται. Δηλαδή τα επόμενα 33 χρόνια θα πρέπει όλα μας τα κτίρια να ανακαινιστούν. Αυτό πρέπει βεβαίως να προγραμματιστεί και θα είναι βασικό στοιχείο της μελλοντική μας κτηριακής στρατηγικής. Τέλος, για την προεκλογική εκστρατεία. Αν κοιτάξουμε τις προηγούμενες προεκλογικές εκστρατείες, το 9, το 14 και τώρα έχουμε τις εκλογές του 19, διαπιστώνουμε ότι αυξάνεται το ποσοστό των δαπανών που δίδεται στα πολιτικά κόμματα. Δηλαδή μειώνεται το ποσοστό στις δαπάνες της ε, θεσμικής προεκλογικής εκστρατείας και δίδονται περισσότερα στα πολιτικά κόμματα για να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους. Οπότε, και φέτος προτείνουμε και είναι συνεπές για την τελική φάση, το 19 δηλαδή, να δώσουμε 17 εκατομμύρια στα πολιτικά κόμματα για να έχουμε μία ε, προεκλογική εκστρατεία για τους candidate τους επικεφαλής των ψηφοδελτίων, σε επαγγελματικό επίπεδο. Θέλουμε να, να ε, διευρύνουμε τις δραστηριότητες για ε, επαγγελματικά διοργανωμένη εκλογική βραδιά, για δυνατότητες ε, συζητήσεων με ε, τους candidate και θέλουμε επίσης να έχουμε μία επιστημονική ε, αναγγελία Τη πρόβλεψη αποτελεσμάτων μισή ώρα μετά το κλείσιμο ε, των εκλογικών τμήματων, ούτω ώστε να το χρησιμοποιήσουν οι εθνικέ τηλεοράσει. Αυτά και ευχαριστώ γιατί έχει περάσει και η ώρα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Γραμματέα. Ξέρω ότι ο κύριος Σασόλη βιάζεται. Ε, δεν θα τον περιμένει η πτήση του. Πέντε έχουν ζητήσει το λόγο. Και θα παρακαλούσα τους διερμηνείς να μας παραχωρήσουν μερικά λεπτά πέραν της εξή... Η κυρία Γκουαρδία Ζαμπάλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους αντιπροέδρους και το Γενικό Γραμματέα που ήρθαν εδώ για να μας δώσουν αυτές τις πληροφορίες. Φυσικά δεν έχουμε ακόμα τα επίσημα έγγραφα γιατί θα πρέπει να περάσουν από το Προεδρείο αλλά παρόλα αυτά λάβαμε σήμερα πολλές πληροφορίες και είναι δύσκολο να αντιδράσουμε έτσι εν μετά από τόσα πολλά στοιχεία που λάβαμε. Νομίζω ότι κατάλαβα ότι η πρόταση που θα, παρουσιάσει, ε, θα παρουσιαστεί θα προβλέπει 3,9% αύξηση. Αυτό 3,9% έχει και το, το 2,3% για τα, τις έκτακτες δαπάνες, ε, λόγω ας πούμε της προεκλογικής εκστρατείας ή όχι. Εάν ναι, για να, σας, να συνδεθώ με τα όσα υποστήριζαν οι σοσιαλιστές είναι να ελέγξουμε τις διοικητικές δαπάνες, δηλαδή να λάβουμε υπόψη μας τον ε, πληθωρισμό ε, βεβαίως, αλλά βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις έκτατες δαπάνες λόγω ε, πέρα, πέρατος της θητείας, της εντολής του Κοινοβουλίου και λόγω προεκλογικής εκστρατείας καθώς και λόγω των προβλημάτων της ασφάλειας. Πάντως, ένα τμήμα των διοικητικών δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούμε να τα ελέγξουμε για να υπάρχει μια ισορροπία με τον προϋπολογισμό. Λοιπόν, τα λεφτά που ξέρουμε για την μετάφραση. Ο Γενικός Γραμματείας έλεγε ότι οι περισσότερες συνεδριάσεις είναι στα αγγλικά. Μερικές φορές υποχρεωτικά όμως, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εκθέσεις που τις λαμβάνουμε ήδη μεταφρασμένες. Ε, αν θέλουμε να τις, μεταφράσουμε, να μεταφράσουμε εντός των προθεσμιών είναι αδύνατον. Για να μπορέσουμε να δουλέψουμε λοιπόν χρειαζόμαστε τα αγγλικά ε, για να παρουσιάσουμε τις τροπολογίες κτλ. Η δουλειά της μετάφρασης και η οργάνωση είναι κάτι πολύ περίπλοκο και είμαστε το μοναδικό θεσμικό όργανο που κάνει, έχει τέτοιο επίπεδο με διερμηνία και μετάφραση. Δεν είναι καθόλου εύκολο κάτι τέτοιο. Ε, μια και κάνουμε μια τόσο σημαντική επένδυση όμως θα πρέπει να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ε, τώρα ξέρω ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα να αρχίσουμε να μιλάμε όλοι αγγλικά. Ε, κύριε Βίγλαντ, μία προτεραιότητα για τους επόμενους προϋπολογισμούς είναι να είμαστε αποτελεσματικοί στις δαπάνες μας. Ο τρόπο που δουλεύουμε στο Κοινοβούλιο πέρασε από πολλέ αλλαγέ και πρέπει να προσαρμοστούμε και προσαρμοστήκαμε. Το να κάνουμε κάποιε δαπάνε και κάποιε επενδύσει είναι λογικό και να αλλάξουν κάποια πράγματα. Είναι ευκαιρία, α πούμε, για να κάνουμε και εξορθολογισμό, α πούμε, και αποτελεσματικότητα κάποιων δομών. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, μα παράλογο. Ζητώ συγγνώμη όμω. για, την, για λόγους ασφάλειας θα πρέπει όλοι να μπαίνουμε με το badge και τα λοιπά. Ε, δεν χρειάζεται τότε να πηγαίνουμε από αίθουσα σε αίθουσα και να, για να υπογράφουμε όλα αυτά τα, τα μητρώα. Είναι μια μπουρδα αυτό το πράγμα. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε ηλεκτρονικά. Είναι, μπορούμε λοιπόν, ε, να, ένας τρόπος για να δουλεύουμε πιο αποτελεσματικά, να τρέχουμε, αντί να τρέχουμε από αίθουσα σε αίθουσα, να το κάνουμε ηλεκτρονικά. Ευχαριστώ. Κύριε Σαλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ρούμπικ, κύριε Σασόλη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη ανάλυση που μας παρουσιάσατε και για όλες ε, τις πληροφορίες που μας δώσατε για τα οικονομικά του Κοινοβουλίου και για το 2019. Έχουμε διαβάσει την έκθεση που έχει υποβληθεί στο Προεδρείο και προέβλεπε ορισμένες προβλέψεις για το 2019. Εκεί βρίσκουμε λεπτομερή στοιχεία για τις ε, πιο σημαντικές εκδηλώσεις που προγραμματίζεται το 2019 το Κοινοβούλιο και συμφωνούμε με την ε, εκτίμηση σε ό,τι αφορά ε, τις οικονομικές συνθήκες και τις προσδοκίες από τις επερχόμενες εκλογές και τα όσα θα προκύψουν από το Brexit. Είπαν και οι συνάδελφοι ότι τα στοιχεία αυτά ε, συνδέονται και με τον, με τον Brexit. Θα είναι ε, το μικρότερο μερίδιο του τομέα 5 από την έναρξη των επιδελταπή. Από την άλλη, ε, σε αιτήσια βάση βλέπουμε τη μεγαλύτερη αύξηση του προπολογισμού του Κοινοβουλίου. Αυτή η αύξηση του 3,9% είναι αιτιολογημένη, τεκμηριώνεται. Όμως ξέρουμε επίσης ότι φτάνουμε στο τέλος της τρέχουσας θητείας και υπάρχει αυξανόμενη πίεση από τις ΜΚΟ και από τα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε προτεραιότητες όπως η οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση, συνοχή. Έχουμε επίσης και διεθνείς δεσμεύσεις, ασφάλεια, άμυνα. Επομένως, είναι προφανές ότι ο Ευρωπαίος φορολογούμενος θα περιμένει από εμά να διοχετεύσουμε κονδύλια σε αυτούς τους τομείς. Δεδομένων όλων αυτών, θα είναι λίγο πιο δύσκολο να αιτιολογήσουμε ορισμένες δαπάνες στον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Και εδώ Έχω κατά νου την ε, υφιστάμενη κοινωνική και πολιτική, οικονομική συγκυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη μιλούμε για προπολογισμούς με βάση ε, τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις. Συνεχώς αυτό λέμε και ξαναλέμε. Θεωρούμε ότι ένας τέτοιος προπολογισμό ε, θα ήταν πιο αποτελεσματικός και θα μας βοηθούσε να εξοικονομήσουμε πόρους. Από την άλλη διαρωτώ με τι θα γίνει με τις επιπρόσθετες υποχρεώσεις μας δεδομένων των προκλήσεων της επόμενης χρονιάς. Ευχαριστώ κύριο Σταράου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάντα χαίρομαι όταν ακούω τις ε, παρατηρήσεις των αντιπροέδρων που πάντα βασίζονται στο, στις σκληρές προσπάθειες ε, του κυρίου Βέλε για την επιβίωση ε, του Κοινοβουλίου. Βεβαίως, όπως είπε και ο κύριος Άλλη, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα τώρα. Το να δούμε δηλαδή όλα τα προβλήματα που έχουμε, όλα τα καθήκοντα, όλες τις υποχρεώσεις μας και από την άλλη πλευρά και να τεκμηριώσουμε τις επιμέρους ε, επιλογές μας ό,τι φορά τις γραμμές προϋπολογισμού και πώς θα πείσουμε το ευρωπαϊκό κοινό, την ε, κοινή γνώμη ότι ήταν απαραίτητη. Μετά από 25 χρόνια το να λέμε ότι το, το κτίριο PHS μετά από 25 χρόνια ε, πάει, πρέπει να το κατεδαφίσουμε δεν ξέρω, από άλλες απόψεις μπορεί να ευσταθεί. Αλλά είναι πολύ δύσκολο για τα μέλη να ε, αιτιολογήσουν προς τα έξω γιατί κάνουμε αυτή την επιλογή. Μας ε, διαβεβαιώσατε ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε τα αγγλικά ως γλώσσα εργασίας. Πολύ καλό αυτό, αλλά σας προειδοποιώ ότι θα είναι παράνομο. Και ο Νάιτζελ Φαράζ θα μας ζητήσει αποζημίωση που χρησιμοποιούμε τη γλώσσα του μετά τον Brexit. Πρέπει να λάβουμε και αυτό υπόψη στον επόμενο προπολογισμό. Το τρίτο που θα ήθελα να επισημάνω. Λοιπόν, ο προπολογισμό για την προεκλογική εκστρατεία. Δεν ξέρω για τους άλλους συναδέλφους, αλλά για μένα αυτό θα είναι αρκετά πολύπλοκο δεν ξέρω δηλαδή πώς να το παρουσιάσω στο λαό μου. Γιατί το θεσμικό όργανο πρέπει να μπει σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Τα πολιτικά κόμματα είναι αυτά που ε, διεξάγουν την ε, προεκλογική εκστρατεία και κατά τη γνώμη μου εκείνοι θα πρέπει ε, να συλλέξουν χρήματα από τα μέλη τους ή από κάπου αλλού, αλλά όχι από τον προπολογισμό. Όμως για την ιστορία. Να σας πω ότι στην Εστονία τα πολιτικά κόμματα δαπανούν 500.000 ευρώ για κάθε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ ξοδεύω 100 φορές λιγότερα. Και τα δανείζομαι από τη μητέρα μου και πρέπει να της τα επιστρέψω. και έτσι είναι και προσωπική υπόθεση του καθένα που θέλει να γίνει πολιτικός εκπρόσωπος να αναλάβει και αυτή την ευθύνη. Δεν ξέρω πώς θα πάνε και τα κληρονομικά σας, ε, κύριε Ταράν. Ποιος? Κύριε Ντανή. Τζάνι. είναι το όνομά μου, πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Μια και είναι ξεμισίδη. Όπως είπαν οι αντιπρόεδροι και ο Γενικός Γραμματέας, το 2019 είναι μια ειδική χρονιά. Υπάρχουν έξοδα, ειδικά εντό αγωγικών, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά συμφωνώ με την ε, κυρία Γκουάρδια Θαβάλ ότι στο γενικό κορβανά των εξόδων του προπολογισμού υπάρχουν γραμμές οι οποίες μπορούν να εξορθολογιστούν για να μειώσουμε το συνολικό όγκο των δαπανών και το συνολικό αυτό κονδύλι, ή μάλλον αυτό το 3,9 που είναι η γενική αύξηση που προτείνεται. Για τα υπόλοιπα σημεία θα τα συζητήσουμε με τους συνεισηγητές. Καταρχάς, ε, τα κονδύλια για την προεκλογική εκστρατεία. Γενικά συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Τάραντ, ότι την προεκλογική εκστρατεία την κάνουν τα κόμματα και όχι τα θεσμικά όργανα για το ποσό των 33 εκατομμυρίων ευρώ. Πρέπει να το ξαναδώ. Δεν βρήκα καμία συγκεκριμένη αναφορά για να καταλάβω πώς στάσατε για την προεκλογική εκστρατεία σε αυτό το νούμερο, ε, ειδικά το 2014. Ή μάλλον, πώς στάσατε τώρα σε αυτό το 33 εκατομμύρια, αφού έχουμε τις ίδιες συνθήκες με το 2014. Επίσης, για αυτή τη γραμμή αν αποφασίσουμε να κάνουμε προεκλογική εκστρατεία, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτή η εκστρατεία θα είναι ουδέτερη. Θα είναι μια εκστρατεία μόνο και μόνο για να πείσουμε του ε, Ευρωπαίου ψηφοφόρου να πάνε να ψηφίσουν στι ευρωεκλογέ. Όχι για να του πείσουμε να ψηφίσουν για το ευρωπαϊκό project. Για αυτό το θέμα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να τηρήσουν συγγύνη ηχθείως. Για τα υπόλοιπα θέματα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε πολύ πιο άνετα με τους συνεισηγητές. Ευχαριστώ τον κύριο Τζάνι, ο κύριος Μάκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Άκουσα πως παρουσιάστηκε ο προπολογισμό και συμφωνώ με τα περισσότερα. Αλλά να σας πω το εξή. Το 2015 οι ευρωβουλευτές έθεσαν στην Κομισιόν 15.200 ερωτήσεις και σιγά σιγά το κατεβάσαμε στις 1.560 ερωτήσεις αυτό είχε ως συνέπεια εξοικονόμηση 5,3 εκατομμύρια. γιατί 105 συνεργάτες του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν έπρεπε να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις. Και ορισμένες ε, ερωτήσεις ε, ήταν εντελώς ακατανόητες. Για παράδειγμα, μια ερώτηση έλεγε πώς θα πρέπει να ασφαλτοστρώσουμε τους δρόμους στην Ιταλία. Τώρα είναι λιγότερες αλλά καλύτερες ερωτήσεις που τίθενται. Προηγουμένως δεν υπήρχε καμία, ε, κανένας έλεγχος, καμία αξιολόγηση. Τι ποιότητα έχουν ερωτήσεις. Το θέμα ήταν απλώς να κάνουν ερωτήσεις οι βουλευτές για να μπορούν να πούνε ότι να κάνω πολλές ερωτήσεις, άρα είμαι δραστήριος. Μία άλλη παρατήρηση. Οι περισσότερες ε, Ε, που προβλέπονται στον προλογισμό προβλέπουν βέβαια και κάποιες πιστώσεις οι οποίες όμως ε, ε, στο τέλος μπορεί να μας οδηγήσει σε εξοικονομήσεις γιατί προβλέπουμε κάποια ποσά για αυξήσεις των μισθών των υπαλλήλων που μετά για διάφορους λόγους δεν πραγματοποιούνται και άρα θα μπορούσαμε να έχουμε προβλέψει αυτήν την, ε, τις λιγότερες δαπάνες και να αξιοποιήσουμε αυτά τα ποσά που θα είχαμε εξοικονομήσει για να, πληρώσουμε, να αποπληρώσουμε ταχύτερα τα κτίρια και να γλιτώσουμε τόκου. Δηλαδή, να καταλάβουμε ότι κάποιε αυτόματες αναπροσαρμογές δεν είναι και τόσο αυτόματε και έτσι θα έχουμε περισσότερα χρήματα για να επενδύσουμε στα κτίρια, στον εξοπλισμό των βουλευτών κτλ. Οπότε, θα ήθελα να μάθω πότε θα εφαρμόσουμε αυτή τη διαδικασία που την έχουμε αποφασίσει δύο φορές και ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μάνκα που υπογραμμίσατε ότι πρέπει να γίνεται βελτιστοποίηση όχι μόνο στον φορολογικό τομέα αλλά και για την ε, σωστή ε, αποτίμηση και αξιολόγηση της εργασίας των βουλευτών, γιατί κάποιοι δείκτες ε, είναι θεωρητικοί. Αύριο θα ψηφίσουμε για τη δημιουργία 49 θέσεων και θέλω να μου πείτε κύριε Γενική Γραμματέα, 49 θέσεις. Ακριβώς ε, για τη στρατηγική ε, για την επικοινωνία κατά την προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, ακούσατε τις παρτίσεις των συναδέλφων πολύ σύντομα γιατί έχουμε πρόβλημα διερμηνίας. Ποιο θα απαντήσει, ο κύριο Βίλαντ. Λοιπόν, λέει ο κύριο Βίλαντ. Κύριε Τάραντ. Όταν δαπανά η Ευρωπαϊκή Ένωση πόρους για να πείσει για παράδειγμα τους πολίτες ότι πρέπει να εξοικονομούν νερό, τότε γιατί να μην μπορεί να πει και στους πολίτες είναι σημαντικό να εκφραστείς μέσω των ε, ευρωεκλογών, να ψηφίσεις, να συμμετάσχεις. Δεν είναι πολιτικό αυτό. Πρέπει να επιτρέπεται στην Ένωση να ε, γνωστοποιήσει ότι γίνονται ευρωεκλογέ. Γιατί να τι διαπιστώσαμε και από τη συμμετοχή των νέων στο δημοψήφισμα στη Βρετανία. Θα ήταν καλύτερα αν είχαν ψηφίσει περισσότεροι νέοι. Αν από πλευρά ε, συντηρητική άποψη ότι ο κύριο Τάραντ είναι εναντίον, τι θα μπορούσα να πω εγώ, θα έλεγα 50 αποχρώσει του πρασίνου. Κυρία Γαρδιαθάβαλ. Τεχνικά επιτεύγματα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας όταν λέτε ότι πρέπει να εξυγχρονιστούν ορισμένα θέματα και για τους ευρωβουλευτές. Αλλά υπάρχουν και θέματα προστασίας δεδομένων και υπάρχουν βουλευτές που λένε εγώ δεν θέλω να με επιτηρούν. Να αναφέρω δύο παραδείγματα. Έχουμε ένα νέο πιλωτικό πρόγραμμα, αυτό για το οποίο σας έχω προσκαλέσει και εσάς κυρία Γαρδιαθάβαλ. Εκεί για παράδειγμα προβλέπετε στο μέλλον να μην έχουμε πλέον ε, ε, ε πολλά κλειδιά επάνω μας, με τα μπάτζ να ανοίγουν τις ε, πόρτες. Άρα ορισμένοι βουλευτές φοβούνται ότι θα μπορούν να διαβάσουν ε, όλοι ποιος, πότε μπαίνουν και πότε βγαίνουν από το γραφείο τους. Και το θέμα είναι επίσης αν κλαπούν για παράδειγμα κάποια κλειδιά, να ξέρουμε πότε κλάπησαν. Και επίσης θα μπορούσαμε με βιομετρικά στοιχεία να μην είναι αναγκαίο να υπογράφουν οι βουλευτές. Αλλά το θέμα είναι πόση αποδοχή υπάρχει. Γι' αυτό κάνουμε ναι, τέτοια πιλωτικά προγράμματα, για να εφαρμόσουμε ε, κάποια συστήματα ξεπερνώντας τους φόβους των βουλευτών. Εγώ όμως πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μέσω πειθού. Και εγώ βεβαίω είμαι διατεθειμένο να προωθήσω αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστώ. Κύριε Γενική Γραμματέα. Ευχαριστώ πολύ. Τέσσερις ερωτήσεις. Πρώτον, ηλεκτρονική υπογραφή. Τεχνικά, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος Βίλαντ, ε, τεχνικά είμαστε πολύ κοντά, αλλά πολιτικά πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις. Άρα πρέπει να ληφθεί η απόφαση του Προεδρείου. Και κατόπιν θα το εφαρμόσουμε. Δεύτερον, Σύγκριση του κόστους των ευρωεκλογών του 2014. Δηλαδή οι δαπάνες αυτής της εκστρατεία του 2014 με, τη, με τις προβλεπόμενες δαπάνες και το 2019 είναι παρόμοια τα ποσά. Αλλά τώρα θα αυξήσουμε τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ούτω ώστε να στηρίξουν τους επικεφαλείς των ψηφοδελτίων τους, τους Spitzenkandidat. Εδώ θα δώσουμε περισσότερα. Είναι σαφές, όπως υπόθηκε, ότι πρέπει να γίνει περισσότερη επικοινωνική δουλειά από τα πολιτικά κόμματα. Ο κύριος Μάνκα είπε ότι διάφοροι δείκτες ε, τελικά είναι κάπως απατηλοί. Υπάρχουν κάποιοι ποσοτικοί δείκτες ε, μέσω των οποίων καθορίζεται ποιος είναι επιμελής ευρωβουλευτής και ποιος λιγότερο και τελικά έχουμε παράλογες καταστάσεις. Κάποιοι δηλαδή υποβάλλουν ένα τεράστιο αριθμό ερωτήσεων. Οπότε μετά στο... Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι να προσαρμόσουμε το, το ανάλογο website για να βασίζεται σε σωστά κριτήρια και όχι απλώς έτσι σε ποσοτικά κριτήρια. Ο κύριος Αρτσουή έθεσε το θέμα των 49 θέσεων. Δεν είναι θέση το οργανόγραμμα. Είναι με συμβόλαια θέσεις για, τον εξωτερικό, για να εργαστούν στα εξωτερικά γραφεία. Δεν αυξάνει τον προπολογισμό, θα είναι πιστώσεις από τις πιστώσεις που προβλέπονται για την προεκλογική εκστρατεία. Το Προεδρείο αποφάσισε ότι τα εξωτερικά γραφεία πρέπει να κάνουν περισσότερη προεκλογική δουλειά ε, μέσω του τύπου, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προτιμάμε να το κάνουμε αυτό μέσω ε, συμβασιούχων παρά μέσω ε, υπεργολαβιών. Ο κύριος Βίμπιχ, 30 δευτερόλεπτα παρακαλώ. Ελπίζω ε, ότι θα μπορούσατε να πείτε το 3,9 να το, να το μειώσουμε, το 3,9 αύξησε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους πάντες για τις προτάσεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ να είμαι καλός εισηγητής για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. επιμένω στην ευχή που εξέφρασα. Ε, έχω εμπιστοσύνη στο Προεδρείο, στο Γενικό Γραμματέα και τα λοιπά, ούτως ώστε να μειωθεί το 3,9%. Αν ε, έχετε υπόψη σας ε, την επόμενη προεκλογική εκστρατεία, ε, καλό θα ήταν να κάνουμε προσπάθειες για να μειωθεί αυτό το νούμερο, το 3,9%. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τους συνεργάτες, ευχαριστώ κυρίως τους διερμηνείς. Γιατί και το μεσημέρι ξεπεράσαμε το όριο που ήταν 12.30 ώρα. Και αύριο μια μεγάλη στιγμή ευτυχίας που θα ξεκινήσει σε 9 η ώρα.